Άρχεται η συνεδρίαση. Ε, χτες ε, το Βρετανικό Κοινοβούλιο εξεφράστη με πολύ μεγάλη πλειοψηφία εναντίον της συμφωνίας η οποία ήταν το αντικείμενο διαπραγμάτευσης τα τελευταία δύο χρόνια με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς θα λάβουμε υπόψη μας το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αυτής με μια κάποια πικρία, αλλά φυσικά θα το σεβαστούμε, διότι είναι η έκφραση της πλειοψηφίας των πολιτικών δυνάμεων που ήσαν παρούσες στην Κάτω Βουλή. Δεν διαφεύγει ότι υπάρχουν πολλές πολιτικές ε, δυνάμεις που καταψήφισαν την συμφωνία, αλλά για διαφορετικούς λόγους άλλοι ανήσυχοι για το backstop, άλλοι ευχόμενοι στενότερη σχέση με την Ένωση στο μέλλον, την διατήρηση της Τελωνιακής Ένωσης. Είναι σαφές ότι είναι νωρίς για να αξιολογήσουμε τις συνέπειες αυτής της ψηφοφορίας. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε όμως τις εξελίξεις και στο Westminster δεν υπάρχουν πλειοψηφίες υπέρ της μίας ή της άλλης υπόθεσης. διαμορφώνονται ουσιαστικά δύο αρνητικές πλειοψηφίες, μία εναντίον της συμφωνίας και η άλλη εναντίον της εξόδου χωρίς συμφωνία, αλλά δεν υπάρχει κάποια θετική πλειοψηφία. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι θα γίνουν προσπάθειες έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια πλειοψηφία υπέρ μιας κοινή λύσης και θα αναμένουμε για να δούμε πώς η Βρετανική κυβέρνηση θα συνεχίσει από εδώ και πέρα. Εμείς από πλευράς μας θέλουμε να επιμείνουμε στις στενές σχέσεις μας με το Ηνωμένο Βασίλειο, εφόσον το επιθυμεί και το ίδιο, και εφόσον αποφασίσει να τροποποιήσει τις κόκκινες γραμμές τις οποίες μας είχε επιβάλει. Εμείς έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στο διαπραγματευτή μας, τον κύριο Μισελ Μπαρνιέ, ο οποίος με ευφυΐα, ικανότητα και σοφία διήφθηνε και κατήφθηνε τις διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι τώρα αν δεν είναι δυνατόν να είμαστε όσο φιλόδεξοι επιθυμούμε, θα οδεύσουμε σε μία έξοδο χωρίς πρώτερη συμφωνία, κάτι το οποίο θα είναι αρνητικό για όλους και το παραδέχονται αυτό όλοι. Παρ' όλα αυτά θα επιταχύνουμε τις προετοιμασίες έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι για μία έξοδο άνευ συμφωνίας. και αυτή είναι και η γραμμή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αυτό το οποίο έχει σημασία είναι να μην αδικήσουμε τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στο Ηνωμένο Βασίλειο και τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου που κατοικούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα πρέπει να υποφέρουν και δεν θα πρέπει να είναι τα πρώτα θύματα μιας άνευ πρώτερης συμφωνίας εξόδου. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με πολύ μεγάλη προσοχή το Ιρλανδικό πρόβλημα δεν θα πρέπει να εγκαταλείψουμε την Ιρλανδία. Θα πρέπει τα σύνορα ανάμεσα στη Βόρεια Ιρλανδία και την δημοκρατία της Ιρλανδίας να είναι ένα ευέλικτο σύνολο σύνορων και να καλύπτει τα συμφέροντα της υγείας, της γεωργίας και της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Θα πρέπει να συνεχίσουμε στα πλαίσια αυτού του καθεστώτος την ενότητα των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που ε, διαμορφώσαμε κατά τη διάρκεια αυτών των μακρόχρονων και δύσκολων διαπραγματεύσεων. Μια ενότητα η οποία δείχνει ότι μπροστά στις δύσκολες καταστάσεις υπάρχει και είμαστε ικανοί να έχουμε μια συνεκτική πολιτική γραμμή. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν τώρα πλέον την συζήτηση με τις δηλώσεις της, ε, του Συμβουλίου και της Επιτροπής εξ του Συμβουλίου. Τον λόγο έχει η Υπουργός, κυρία Μελάνια Τσότ. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, τον Νοέμβριο πέρσι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε την Συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρατόμ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Συμβούλιο ενέκρινε επίσης την πολιτική δήλωση η οποία έθετε το πλαίσιο για τις μελλοντικές σχέσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ηνωμένο Βασίλειο και επανέλαβε την αποφασιστικότητα της Ένωσης να έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο στο μέλλον. Αυτό το αποτέλεσμα δεν θα ήταν δυνατόν χωρίς την ενότητα και την υπευθυνότητα μεταξύ των 27 κρατών μελών όπως και μεταξύ των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα Αφού μάθαμε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, δεν μπορούμε παρά να λυπηθούμε για αυτήν, το, αυτό το αποτέλεσμα και θα έχουμε μια άτακτη έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου. Μάλλον ένα τέτοιο σενάριο θα έχει σοβαρές επιπτώσεις για όλους μας, αλλά κυρίως για το Ηνωμένο Βασίλειο. Με τις τα αποτελέσματα θα πρέπει ε, να κάνουμε έκκληση για μεγαλύτερη ενότητα και υπευθυνότητα μεταξύ των κρατών μελών και των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω των πολλών ε, δισταμένων ε, σημάτων που είχαμε πριν από την συζήτηση που οδήγησε στην ψηφοφορία σε όλο το φάσμα το πολιτικό του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι δύσκολο να ξεχωρίσουμε μια εξήγηση γι' αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό το αποτέλεσμα βεβαίως δεν είναι το τέλος του παιχνιδιού, ενώ έχουμε ε, τα ορισμένα μέτρα δεν έχουμε θέμα επαναδιαπραγμάτευσης. Θα πρέπει να δράσουμε όταν το Ηνωμένο Βασίλειο θα έχει διευκρινίσει τι σημαίνει το αποτέλεσμα αυτό για τη διαδικασία κύρωσης και ποιες θα είναι τα επόμενα μέτρα. Εν τω μεταξύ, όπως έκανα έκκληση και έκανε έκκληση το Συμβούλιο στην πρόσκληση στην Κομισιό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα. Εξακολουθούμε την διαδικασία κύρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άποψη αυτή χαίρομαι που μπορώ να αναφέρω ότι την περασμένη εβδομάδα ήδη το Συμβούλιο υιοθέτησε την απόφαση για την υπογραφή της συμφωνίας και ενέκρινε την πρόταση αυτή όπως και ε, το αίτημα για την συγκατάθεση του Κοινοβουλίου. Η υπευθυνότητα για να εξασφαλίσουμε την κύρωση παραμένει ε, στα χέρια της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου. Η αποφασιστικότητά μας να συνεχίσουμε θα έπρεπε να στηρίξει το, την κυβέρνηση για να εκπληρώσει το τελικό αποτέλεσμα ως προς το χρόνο και το περιεχόμενο. Παρόλα αυτά δεν είναι βέβαιο το αποτέλεσμα. Εμείς συνεπώς πρέπει να συνεχίσουμε την προετοιμασία μας για όλες τα ενδεχόμενα ακόμα ε, και για μη συμφωνία. Δεν θέλουμε μια τέτοια κατάσταση, αλλά θα πρέπει να προετοιμαστούμε δεόντως αν υπάρξει μια τέτοια λύση. Η ετοιμότητα και ε, το έκτακτο σχέδιο ανάγκης ε, θα πρέπει να κατέχουν μεγαλύτερη σημασία εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση και σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να προετοιμαστούμε. Αυτό σημαίνει πρόσθετη νομοθετική εργασία σε αυτήν την, τελευταία φάση, αλλά έχουμε εμπιστοσύνη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ανταποκριθεί στην πρόκληση όλων των ενδιαφερομένων. Το Προεδρείο με τη δική σας συνεργασία πάντως είναι αποφασισμένο να διευκολύνει την έγκριση των μέτρων εκτακτής ανάγκης εν ευθέτω χρόνο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Το λόγο έχει ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Φραντς Τίμερμανς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ψηφοφορία στο βράδυ στη Βουλή των Κοινοτήτων ήταν σαφής, απορρίφθηκε η συμφωνία. η Επιτροπή λυπάται ιδιαίτερα για αυτό το αποτέλεσμα, γιατί θεωρούμε ότι ήταν ε, η καλύτερη δυνατή κατάληξη. Είχαμε δύο πλευρές που διαπραγματεύονταν, ο καθένας προσπαθούσε να εξυπηρετήσει τα συμφέροντά του. Ο Μισελ Μπανιέ από πλευρά τη Επιτροπή έκανε μια καταπληκτική δουλειά για να διαπραγματευτεί από πλευρά των 27. Η Βρετανική κυβέρνηση βεβαίω διαπραγματεύτηκε από πλευρά του Ηνωμένου Βασιλείου. Και θεωρούμε ότι το αποτέλεσμα αυτή τη διαπραγμάτευση οδήγησε σε μια συμφωνία αποχώρηση που έκανε τη μικρότερη δυνατή ζημιά. Και να μην έχουμε καμία αυταπάτη το Brexit θα θίξει το Ηνωμένο Βασίλειο, θα θίξει και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ως πολιτική πρέπει να περιορίσουμε την ζημία αυτή στο μέγιστο. Και θεωρούμε ότι η συμφωνία αποχώρησης μας βοήθησε. Θα βοηθούσε προς αυτήν την κατεύθυνση. Βέβαια τώρα εμείς δεν ξέρουμε τι είδους Brexit θα έχουμε. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στη Βουλή των Κοινοτήτων, να δούμε ποια θα είναι η θέση της Βρετανικής κυβέρνησης του Βρετανικού Κοινοβουλίου και θα δούμε μετά τι θα κάνουμε. Αλλά έχουμε υποχρέωση να είμαστε προετοιμασμένοι για οποιαδήποτε δυνατή κατάληξη. Ακόμη και μία άτακτη έξοδο σε περίπτωση έλλειψη συμφωνία που θα έχει πολύ σοβαρέ επιπτώσει και για το Ηνωμένο Βασίλειο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι προετοιμασμένη για να αντιδράσουμε όσο καλύτερα γίνεται σε οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Όπως είπε και εκπρόσωπος του Συμβουλίου, θα συνεχίσουμε τη διαδικασία επικύρωσης της Συμφωνίας Αποχώρησης, εφόσον συμφωνήθηκε. Είναι, κατά τη γνώμη μας, η καλύτερη κατάληξη για να υπάρξει συντεταγμένη αποχώρηση. Και να αναφέρω κάτι, μια παράθεση από το C.S. Lewis. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε και να αλλάξουμε την αρχή, αλλά μπορούμε να ξεκινήσουμε από εδώ που ε, είμαστε και να αλλάξουμε την κατάληξη. Ευχαριστώ πολύ. Τον λόγο έχει τώρα ο υπεύθυνος διαπραγματευτής από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του συνόλου της Ένωσης, ο κ. Μισελ Μπαρνιέ. Ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, μέλη του Κοινοβουλίου, κύριε Αντιπρόεδρε, κυρία Υπουργέ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της την ψηφοφορία στην Κάτω Βουλή που έγινε χθε το απόγευμα και όπως είπε ο πρώτος αντιπρόεδρος, ο κύριος Τίμερμανς, η Κάτω Βουλή ψήφισε χθε με μια ξεκάθαρη πλειοψηφία, ισχυρή πλειοψηφία, εναντίον της συμφωνίας την οποία είχαμε συμφωνήσει, συμβούλιο με την Βρετανική κυβέρνηση, ήδη από τον μήνα Νοέμβριο, και την οποία σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχατε δεχθεί ευνοϊκά. Βέβαια τη στιγμή αυτή είναι πρόωρο να αξιολογήσουμε τις συνέπειες της ψήφου αυτής. Εμείς σεβόμεθα την ψήφο αυτή και θα συνεχίσουμε να σεβόμεθα την δημοκρατική συζήτηση στο Ηνωμένο Βασίλειο και δεν θα ήθελα τώρα να κάνω προφητείες για τα διάφορα σενάρια. Αυτό το οποίο έδειξε η χθεσινή ψηφοφορία είναι ότι οι πολιτικές συνθήκες και προϋποθέσεις για την επικύρωση της συμφωνίας δεν υπάρχουν στο Λονδίνο. Ε, εκφράζουμε τη λύπη μας για την ψηφοφορία αυτή, για το αποτέλεσμα αυτό, όπως το είπε και ο πρόεδρος Γιούνκερ. Αυτό είναι κάτι το οποίο συνδέεται και με την τεράστια προσπάθεια την οποία έχουμε κάνει μαζί σας και με την υπεύθυνη ομάδα ε, για το Brexit εδώ και δύο χρόνια και τη συζήτηση με, το βετανικό, με τη Βρετανική πλευρά, τη Βρετανική κυβέρνηση, η οποία βασίστηκε στις κόκκινες γραμμές της ίδιας της κυβέρνησης αυτής. Λυπούμεθα λοιπόν για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αυτής. Θυμίζω ότι εμείς δημιουργήσαμε από κοινού με τους Βρετανούς, με τη Βρετανική κυβέρνηση, την συμφωνία αποχώρησης επί μιας αντικειμενικής βάσεως, λαμβάνοντας υπόψη ε, την κατανομή των συμφερόντων για να μην υπάρχουν σύνορα στην Ιρλανδία, σεβόμεθη φυσικά την επιθυμία των Βρετανών να διατηρήσουν την εθνική τους κυριαρχία στο σύνολο του εδάφους τους και συνεργαζόμενοι ε, με την, Ευρωπαϊκή, με την Βρετανική κυβέρνηση έτσι ώστε να διαμορφώσουμε το πλαίσιο μιας μελλοντική λύσεως η οποία να μην είναι μακρινή στο μέλλον και ταυτόχρονα όμως να είναι και αρκετά φιλόδοξη όσο θα το επιτρέψουν τουλάχιστον οι Βρετανικές κόκκινες γραμμές. Διαπιστώνουμε κυρίες και κύριοι ακούγοντας τις δημόσιες δηλώσεις ότι οι βουλευτές της Κάτω Βουλής οι οποίοι καταψήφισαν την συμφωνία που έγινε αντικείμενο διαπραγμάτευσης όπως το θύμισε και ο πρόεδρός σας το έκαναν για εντελώς διαφορετικούς λόγους. Πολλές φορές πλήρως αντιτιθέμενους και αντιφατικούς ψηφοφορία αυτή, αντικειμενικά λοιπόν, δεν είναι η έκφραση μιας λεγόμενης θετικής πλειοψηφίας, η οποία θα έθετε μια εναλλακτική πρόταση στη συμφωνία που έχουμε ήδη καταθέσει. Και στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε και πολύ σωστά ο κύριος Τίμερμανς, ανήκει στις Βρετανικές αρχές να αξιολογήσουν την ψηφοφορία αυτή και η Βρετανική κυβέρνηση θα πρέπει να μας πει το πώς θέλει να συνεχίσει από εδώ και πέρα προς μια διατεταγμένη αποχώρηση στις 29 Μαρτίου όπως το υπενθύμησε και ο Ντόναλτ Τάσκ χτες το βράδυ ο πρόεδρος του Συμβουλίου. Κυρίες και κύριοι, αντίθετα από αυτά τα οποία ακούστηκαν τις τελευταίες εβδομάδες και τις τελευταίες ημέρες, η συμφωνία στην οποία έχουμε καταλήξει με τη Βρετανική κυβέρνηση, μια συμφωνία 600 σελίδων, είναι μια καλή συμφωνία είναι φυσικά αποτέλεσμα ενός συμβιβασμού, αλλά είναι ο καλύτερος δυνατός συμβιβασμός. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να εργαζόμαστε με αντικειμενικότητα. Η συμφωνία αυτή παρέχει νομική ασφάλεια, ασφάλεια δικαίου, εκεί όπου το Brexit δημιουργεί ανασφάλεια όπως και κάθε διαζύγιο. Ασφάλεια για τους πολίτες και τους Βρετανούς πολίτες και τους πολίτες των υπόλοιπων 27 χωρών, των οποίων τα δικαιώματα γίνονται αντικείμενο εγγύησης διαρκούς. Αυτή ήταν η βασική μας προτεραιότητα, αυτή ήταν η δική σας προτεραιότητα στο Κοινοβούλιο και η προστασία των δικαιωμάτων αυτών θα παραμείνει η προτεραιότητά μας ανεξαρτήτως των εξελίξεων ασφάλεια επίσης και για τους επιχειρηματίες και σε επίπεδο ιδιωτικό και σε επίπεδο δημόσιο. Όσοι χρησιμοποιούν τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και τροφοδοτούνται από αυτόν, είτε είναι Βρετανοί είτε από τις υπόλοιπες 27 χώρες, όλα αυτά τα προγράμματα γίνονται σεβαστά με βάση αυτή τη συμφωνία. Ασφάλεια και σταθερότητα για τη δημοκρατία της Ιρλανδίας και τη Βόρεια Ιρλανδία, όπου η επιστροφή των σκληρών συνόρων μπορούμε να την αποτρέψουμε με μια ευέλικτη λύση που θα επιτρέψει και θα σέβεται το σεβασμό της κυριαρχίας του Ηνωμένου Βασιλείου και τις ελευθερίες της ενιαίας αγοράς στα πλαίσια της συμφωνίας του Μπέλφαστ, της συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής. Και γι' αυτό ακριβώς εμείς το backstop το οποίο συμφωνήσαμε με το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να παραμείνει ένα αξιόπιστο backstop Πρέπει ένα πραγματικά αξιόπιο backstop, επαναλαμβάνει στην Αγγλική ο κύριος Μπαρνιέ. Δημιουργεί ασφάλεια για τις επιχειρήσεις και για τις δημόσιες διοικήσεις που θα έχουν στη διάθεσή τους ε, μια μεταβατική περίοδο ε, τον οποίο η μοναδική βάση βέβαια λειτουργίας θα είναι η ενδιάμεση συμφωνία η οποία θα τους δώσει χρόνο για να προετοιμαστούν και να προσαρμοστούν. Η συμβιβαστική αυτή πρόταση μας δίνει επίσης μέσω αυτή τη μεταβατική περίοδου τον χρόνο ο οποίος απαιτείται για να διαπραγματευτούμε τις μελλοντικέ μας σχέσεις επί τη βάση των πολιτικών συμφωνιών στις οποίες καταλήξαμε Ένωση και Βρετανική κυβέρνηση και κάποιες αξιολογήσεις κοινέ πολιτικές οι οποίες αφήνουν ανοιχτές τις επιλογές σεβόμενοι όμως τις βασικές αρχές των ΜΕΝ και των ΔΕ. Όπως και να έχουν τα πράγματα, η επικύρωση συγγνώμη, αυτής της συμφωνίας είναι απαραίτητη, είναι προϋπόθεση για τη δημιουργία της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ μας στα πλαίσια της προοπτικής της δεύτερης διαπραγμάτευσης η οποία θα πρέπει να ξεκινήσει το ταχύτερο δυνατόν σχετικά με τις μελλοντικέ μας σχέσεις. Για αυτές τις σχέσεις, τις μελλοντικέ σχέσεις, αυτό που είναι το πιο σημαντικό για το μέλλον και του Ηνωμένου Βασιλείου και της Υπήρου μας, να θυμίσω ότι το κοινοβούλιο σας, το Συμβούλιο ομόφωνα, πάντα έλεγαν και λέγουν ότι εάν το Ηνωμένο Βασίλειο αποφασίσει να αλλάξει τις κόκκινες γραμμές του στο μέλλον και αν το Ηνωμένο Βασίλειο κάνει την επιλογή να σταθεί πιο φιλόδοξα και να ξεπεράσει μια απλή συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών που και αυτή είναι βέβαια σημαντική τότε σε αυτή την περίπτωση η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι πάντα δεκτική έτσι ώστε να συνοδεύσει τις εξελίξεις αυτές και να ανταποκριθεί σε αυτές τις εξελίξεις θετικά. Αναφερόμενο στις μελλοντικές σχέσεις, δεν αναφέρομαι στις οικονομικές εμπορικές σχέσεις, στις συναλλαγές που είναι φυσικά τόσο σημαντικές για την ανάπτυξη και τη θέση απασχόλησης σε μας. Αναφέρομαι και σε τομιακές συνεργασίες στις οποίες εμένουν πολλές κοινοβουλευτικέ ε, ε, επιτροπές σας, πανεπιστήμια, έρευνα, αλληλεία, αερομεταφορές, μεταφορές γενικότερα, συνεργασία σε επίπεδο αστυνομικής, ε, αστυνομικού επίπεδου, δικαστικού επίπεδου, πολύ σημαντικό μετά τον Brexit, η σταθερότητα της Υπήρου μας, η ασφάλεια της Υπήρου μας, η ασφάλεια του Ηνωμένου Βασιλείου, μεγάλης χώρας, μέλους του Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών, χώρα φίλη, χώρα σύμμαχος, χώρα που θα παραμείνει σημαντικός εταίρος σε ό,τι έχει σχέση με την εξωτερική πολιτική, με την ανάπτυξη της συνεργασίας στον τομέα της άμυνας. Κυρίες και κύριοι, έχουμε διεξάγει τους τελευταίους 18 μήνες μια συλλογική προσπάθεια. Η συλλογική προσπάθεια αυτή έχει επικυρωθεί σε κάθε κομβική στιγμή από την Βρετανική κυβέρνηση, από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και από εσάς τους ιδίους. Νομίζω ότι θα υπάρξει λύση σε αυτό το αδιέξοδο, αλλά δεν θα υπάρξει λύση αυτή όσο δεν διευκρονιστούν οι όροι της εξόδου και δεν κατοχυρωθούν από μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία στο Ηνωμένο Βασίλειο και γι' αυτό τα επόμενα στάδια θα πρέπει πλέον να καθοριστούν πλήρως από πλευρά της Βρετανικής κυβέρνησης. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ένα διατεταγμένο Brexit παραμένει η απόλυτη προτεραιότητά μας για τις επόμενες εβδομάδες. Όμως, τη στιγμή που σας ομιλώ, κανένα σενάριο δεν μπορεί να αποκλειστεί. Και αυτό ισχύει επίσης και για το σενάριο το οποίο πάντα θελήσαμε να αποτρέψουμε το λεγόμενο no deal, μη συμφωνία. Είμαστε στις 10, την 16η Ιανουαρίου, 10 εβδομάδες μόνο πριν το τέλος του Μαρτίου, δηλαδή τη στιγμή που επέλεξε η ίδια η Βετανική κυβέρνηση, επέλεξε η ίδια Βετανική κυβέρνηση έτσι ώστε να καταστεί τρίτη χώρα. Δέκα εβδομάδες πριν λοιπόν ποτέ ο κίνδυνος ενός no deal δεν ήταν τόσο υψηλός. Εμείς σαν βασικό στόχο έχουμε να αποφύγουμε ένα τέτοιο σενάριο. Έχουμε όμως την ευθύνη να βλέπουμε τα πράγματα ξεκάθαρα. Και γι' αυτό από δικής μας πλευράς θα εντατικοποιήσουμε τις προσπάθειες για να είμαστε προετοιμασμένοι και για αυτό το σενάριο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου, εδώ και πολλούς μήνες συνεργαζόμενοι με τα κράτη-μέλη και μαζί σας, ε, πρέπει να επιταχύνουμε τις προσπάθειες αυτές σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκομένους μέσα σε σύντομες χρονικές προθεσμίες μπορεί να κληθείτε να πάρετε μέτρα ε, κατεπήγοντα έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες αυτού του σενάριου του απευκταίου. Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας. Η πεποίθησή μας, όπως το υπενθύμησε ο Αντιπρόεδρος Τίμερμανς, είναι ότι η συμβιβαστική λύση την οποία προτείναμε μετά από 18 μήνες διαπραγματεύσεων με τη Βρετανική κυβέρνηση είναι η καλύτερη δυνατή συμβιβαστική λύση. Είναι καρπός επικοδομητικών προσπαθειών από πλευράς των δύο, μερών καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Είναι επίσης αποτέλεσμα μιας επικοδομητικής στάσης δικής μας, δικής μου, στα πλαίσια ηρεμίας, γαλήνης, διαλόγου και διαφάνεια. Τώρα η Βρετανική πλευρά θα πρέπει να διευκρινίσει τον τρόπο με τον οποίο θέλει να προχωρήσει από εδώ και πέρα για να περάσουμε στην απόσυρση τη διατεταγμένη την οποία έχει επιθυμήσει και πως πέραν αυτής της αποχωρήσεως θα οικοδομήσει μαζί μας μια εταιρική σχέση διαρκή και αποτελεσματική. Κύριε Μπαρνιέ, εγώ μπορώ ήδη να προβλέψω ότι θα έχετε την εμπιστοσύνη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά ήταν σαφή και μέσω του χειροκροτήματο. Ε, Σα ευχαριστώ πολύ. Και θέλω να ευχαριστήσω και την ομάδα εργασία μα που συνεργάστηκε πολύ στενά με τον κύριο Μπαρνιέ για να έχουμε την ε, βέλτιστη λύση. Και ιδιαίτερα τον επικεφαλή τη ε, ομάδα του Κοινοβουλίου, τον κύριο Φερχόφστατ, αλλά και τα άλλα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εργάστηκαν τόσο σκληρά για το θέμα αυτό. Και τώρα έχουμε τις ομιλίες. Πρώτα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέιμπερ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Μισελ, κύριε Αντιπρόεδρε, Προεδρία του Συμβουλίου, αγαπητοί συνάδελφοι. Τέσσερι σύντομε παρατηρήσει. Πρώτα απ' όλα είμαι περήφανο ω Ευρωπαίο. Θυμάμαι αυτά που είχαν υποθεί πριν από δυόμιση χρόνια. Πολλοί έλεγαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ε, αντιμετωπίσει ένα φαινόμενο ντόμινο και άλλοι θα σκοθούν να φύγουν. Θυμηθείτε όμως τώρα τι έγινε. Η, τα 27 κράτη-μέλη είναι ενωμένα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στηρίζει τις θέσεις μας, όλοι ξέρουμε τι θέλουμε. Νομίζω ότι ε, όλοι στην Ευρώπη αντιλαμβάνονται την ισχύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα οι Ιρλανδοί φίλοι μας. Μπορούμε να είμαστε περήφανοι για αυτό που επιτύχαμε τους τελευταίους μήνες, χάρη στο Μισελ, χάρη στην εργασία του και στην δέσμευση του Jean-Claude Όλα αυτά είναι πολύ καλά. Δεύτερον, 28 κυβερνήσεις ευβεβαίωσαν σε τη συνθήκη και τα τρία θεσμικά όργανα είπαν αυτή είναι μια καλή συμφωνία. Και υπάρχει όμως τώρα το όχι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με σαφή πλειοψηφία Άρα οι Βρετανοί φίλοι μας θα πρέπει να κάνουν τα περαιτέρω βήματα. Υπάρχουν αυτοί που θέλουν να αποχωρήσουν ε, χωρίς ε, συμφωνία, υπάρχουν αυτοί που θέλουν ε, σε τα συν, αυτοί που θέλουν να παραμείνουν. Πείτε μας παρακαλώ, τι θέλετε να επιτύχετε. Δώστε μας μια σαφή κατεύθυνση. Και η Ευρώπη είναι διατεθειμένη να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τρίτον, ξανασκεφτείτε τους στόχους μας. Ε, θα είναι δύσκολη η πολιτική κατάσταση στο μέλλον. Είχαμε σαφείς αρχές όταν ξεκινήσαμε τη συζήτηση. Για μένα, για παράδειγμα, η ιδέα της ενιαίας αγοράς και της ελεύθερης κυκλοφορίας των Ευρωπαίων στην Ήπειρο, ότι μπορούν να αποφασίσουν πού θέλουν να διαμένουν. Αυτό είναι ένα τεράστιο επίτευγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και, όπως και στο παρελθόν, θα υπερασπιστώ αυτή την αρχή. Οποιοδήποτε το αποτέλεσμα της διαδικασίας εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου. Και υπάρχουν και άλλα θέματα δεν θέλουμε να υπάρχουν έλεγχοι στην, στα σύνορα της Ιρλανδίας ή να διατηρηθούν τα δικαιώματα των ε, πολιτών. Δεν βλέπω να υπάρχει καμία δυνατότητα ελιγμών για αναδιαπραγμάτευση. Αν έχουν ε, περαιτέρω αιτήματα, τότε έχουμε και εμείς ε, το δικαίωμα να προβάλλουμε περαιτέρω αιτήματα και όλα θα ξαναρχίσουν. Θα ξανανοίξει η συζήτηση. Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν υπάρχει καμία δυνατότητα αναδιαπραγμάτευσης. Και τέλος, ταξιδεύω παντού στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή ως υποψήφιος, όπως ε, και πολλοί από εσά. Και δεν βλέπω κανένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θεωρεί ότι η Βρετανική προσέγγιση είναι ευφύη. Κανείς δεν μου λέει κάτι τέτοιο. Οι πολίτες της Ένωσης μου λένε ότι βλέπουν ε, πολιτικό χάο, βλέπουν οικονομική αβεβαιότητα. Γι' αυτό το κύριο μήνυμά μα στην προεκλογική εκστρατεία είναι μην ακούτε του εθνικιστέ, του εγωιστέ. Είναι ψεύτε. Πολύ καλύτερα να μεταρρυθμίσουμε την Ένωση παρά να φεύγει κανεί ή να επιχειρεί να καταστρέψει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριο Ρομπέρτο Γκουαλτιέρη, εξ ονόματο τη Προεδρευτική Συμμαχία Σοσιαλιστών. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μετά από δύο μήνες αναβολών γνωρίζουμε τη θέση πλέον της, της Βρετανικής Βουλής. Μια τεράστια πλειοψηφία καταψήφισε την Συμφωνία Απόσυρσης και την πολιτική δήλωση που τη συνοδεύει. Είναι μια ιστορική ήττα για τη Βρετανική κυβέρνηση και την Πρωθυπουργό Μέη. Γνωρίζουμε τώρα αυτό που δεν θέλει το Βρετανικό Κοινοβούλιο αλλά 70 μέρες πριν από την τελική ημερομηνία δεν ξέρουμε το τι θέλει το Βρετανικό Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο ξεκαθάρισε την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα αρνηθεί ένα σενάριο μη συμφωνίας, ένα no deal, γιατί αυτό είναι το χειρότερο σενάριο για όλους και για το ίδιο το Ηνωμένο Βασίλειο κυρίως. Εμείς επαναλαμβάνουμε λοιπόν την δήλωσή μας αυτή, δεν αποσύρουμε, δεν ε, δεν θέλουμε να καταστήσουμε πιο χαλαρή τη συμφωνία αυτή, θέλουμε να προστατεύσουμε την κατάσταση στην Ιρλανδία και στη Βόρεια Ιρλανδία, θέλουμε να αποφύγουμε τα σκληρά σύνορα, θέλουμε να διατηρήσουμε την ενιαία αγορά, όλα αυτά δεν τα διαπραγματευόμεθα. Το να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η βασική μας προτεραιότητα και η αδίποτε λύση που απειλεί τα δικαιώματα αυτά δεν θα γίνει δεκτή η ασφάλεια των συνόρων είναι εξίσου σημαντική με τα επίπεδα τα κοινωνικά, τα οικονομικά, τα φορολογικά, την ισορροπία δικαιωμάτων και καθηκόντων, όλα αυτά σε καμία περίπτωση δεν θα αμφισβητηθούν. Και δεν θα υποκύψουμε επίσης σε αδίποτε πρόκληση για διμερείς λύσεις, η οποία δεν θα είναι ωφέλιμη για τις δύο πλευρές η ενότητα ανάμεσα στα όργανα, η ενότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα πλαίσια της στήριξης του κύριου διαπραγματευτή μας ήταν και θα παραμείνει η βασική μας ισχύς. Ε, είμαστε ενωμένοι και θα συνεχίσουμε να σε υποστηρίζουμε, Μισελ. Πού θα πάμε από εδώ και πέρα. Απαιτείται μια θετική πλειοψηφία από πλευράς Βρετανών. Απαιτείται ένας ξεκάθαρος ορίζοντας και μια ικανότητα να καταλήξουμε σε λύσεις. Η ψηφοφορία χθε απέδειξε ότι κάτι τέτοιο δεν υπάρχει σήμερα. Η υποστήριξη ε, από την πλειοψηφία λοιπόν της κυβέρνησης αυτής μπορεί σήμερα να την διατηρήσει στην εξουσία στην απογευματινή ψηφοφορία αλλά δεν δίνει την απάντηση στο σημαντικό ερώτημα ε, ή θα υπάρξει μια θετική πλειοψηφία υπέρ του Brexit και θα διαμορφωθεί στην Βρετανική Βουλή ή θα πρέπει να ξαναυπάρξει ένα δημοψήφισμα. Αν το Ηνωμένο Βασίλειο θέλει να αλλάξει τις ε, ερυθρές γραμμές της, ε, τότε εμείς θα παραμείνουμε ε, σε στενή σχέση μαζί του. Εμείς βέβαια τις γραμμές αυτές προσπαθήσαμε να τις συζητήσουμε, αλλά δεν κατέστη δυνατό να συμφωνήσουμε σε όλες. Νομίζω ότι μπορεί να επιδειχθεί ρεαλισμός και από τις δύο πλευρές και θα πρέπει με επικοδομητικό τρόπο να σεβαστούμε τις κατευθυντήριες γραμμές μας και τις ε, κόκκινες γραμμές μας που έχουμε διαμορφώσει από το παρελθόν. Σεβόμεθα το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, αλλά θεωρούμε το Brexit ένα ιστορικό λάθος, το οποίο δυστυχώς θα αντιμετωπίσει με αρνητικό τρόπο τον Βρετανικό λαό. Ε, το άρθρο 50 δεν μπορεί να αλλάξει έτσι όπως είναι τώρα και αν ε, δεν μπορούμε στη Βρετανική Βουλή να βρούνε μία λύση από εδώ και πέρα, τότε ίσως θα πρέπει να υπάρξει δυνατότητα είτε νέων εκλογών είτε νέου δημοψηφίσματος. Η πολιτική μας ομάδα είναι ξεκάθαρη ότι αν μία διεύρυνση του άρθρου 50 είναι κάτι το οποίο απαιτείται έτσι ώστε να δοθεί χρόνος για τις δύο αυτές επιλογές, για οποιαδήποτε από τις δύο αυτές επιλογές, φυσικά θα συμφωνήσουμε. Αλλά μια παράταση θα πρέπει να είναι τεκμηριωμένη και όχι για να χάσουμε ακόμα περισσότερο χρόνο. Το Brexit είναι σε αδιέξοδο. Τώρα ε, θα πρέπει το Ηνωμένο Βασίλειο να δείξει υπεύθυνη η ηγετική θέση, να ξεκαθαρίσει τις επιθυμίες της και να προσπαθήσει να οδηγήσει τη χώρα εκτός των δυσκολιών. Εμείς θα παραμείνουμε αξιόπιστοι εταίροι, θα παραμείνουμε επικοδομητικοί εταίροι, εργαζόμενοι υπέρ των συμφερόντων των ευρωπαϊκών λαών. Από πλευρά των Ευρωπαίων Συντηρητικών, ο κύριος Κάμαλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Τίμερμανς. Καταρχά να ευχαριστήσω και τον κύριο Μπαρνιέ και τον κύριο Τίμερμανς για τι μετρημένε ομιλίε του. Νομίζω ότι ήταν πολύ σωστοί και δεν νομίζω ότι μπορεί να διαμαρτυρηθεί κανεί ε, για αυτά που είπαν. Να σα ε, μιλήσω ω κάποιο που παρατήρησε τη συζήτηση για την συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου από τι δύο πλευρέ ε, τη μάχη, Έχω μιλήσει με πολλά άτομα και από τι δύο πλευρέ των διαπραγματεύσεων και προτείναμε λύσεις για να ξεπεράσουμε κάποιε δυσκολίε και ω επικεφαλή τη ομάδα μου. Δεν ε, σας είπα μόνο με τι είμαστε αντίθετοι, αλλά πρότεινα και εναλλακτικέ λύσεις. Από τότε που έγινε ευρωβουλευτής, κάτι που μου έκανε εντύπωση στι σχέσει Ηνωμένου Βασιλείου Ευρωπαϊκή είναι πόσο διαφορετικά αντιμετωπίζετε από τι δύο πλευρέ τη μάχη. Πολλοί πιστεύουν στο μοντέλο ε, πολιτική ενοποίηση μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ενώ στα τελευταία 40 χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο η πολιτική τάξη ε, παρουσιάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση ως χώρο εμπορίου. Δεν αναφέρονται ή υποτιμούν την πολιτική ενοποίηση. Το γεγονό ότι η πολιτική έχει να κάνει με το πώ αντιλαμβάνονται οι συμπολίτε, έχει να κάνει επίση με το πώ αντιμετωπίζεται από τι δύο πλευρέ η αποχώρηση. Από ε, αυτή την πλευρά είπε σαφώ η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλουν να τιμωρήσουν κανένα, αλλά Όποιο ε, αποχωρεί δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται όπω αντιμετωπίζονται τα μέλη. Είχατε μια ε, σκληρή στάση διαπραγματεύσει. Όχι μόνο γιατί είναι καλό αυτό για οποιοδήποτε διαπραγματευτεί, αλλά ούτω ώστε οποιαδήποτε συμφωνία να είναι αντικίνητρο για οποιοδήποτε άλλη χώρα θα μπορούσε να σκεφτεί ότι θέλει να αποχωρήσει. Οι περισσότεροι εδώ στο Κοινοβούλιο χαίρονται που οι στόχοι αυτοί επετεύχθησαν. Αλλά μου τονίζουν ότι έγιναν και συμβιβασμοί στην πορεία. Ορισμένοι ανησυχούν ότι το backstop μπορεί να δώσει ε, ένα αθέμητο προτέρημα στις βρετανικές επιχειρήσεις που θα έχουν πρόσβαση στην ενιαία αγορά. Άλλοι θεωρούν ότι μπορεί να μειώσει τη δυνατότητα στο μέλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνάψει συμφωνίες και μου είπαν ότι ελπίζουν δεν θα χρειαστεί το backstop. Το είπαν πολλοί ομιλητέ εδώ. Αλλά στο Westminster οι αντίπαλοι αυτή ε, τη συμφωνία το βλέπουν πολύ διαφορετικά. Για άλλη μια φορά είναι πολύ μεγάλο το χάσμα στην, ε, στο πώ αντιλαμβάνονται οι δύο πλευρέ. Θεωρούν ότι είναι μια ε, συμφωνία αποχώρηση με νομικέ υποχρεώσει που θεωρούν ότι μπορούν να του εμπλέξει σε μια τελειωνιακή ένωση για πάντα. Ορισμένοι υπεύθυνοι τη Κομισιόν είπαν ότι η τελειωνιακή ένωση θα είναι η βάση για τη μελλοντική σχέση και θεωρούν ότι το κείμενο αυτή τη συμφωνίας δεν περιέχει την υποχρέωση να περάσουμε σύντομα σε ε, συμφωνία ελευθέρου εμπορίου. Λένε ότι ναι μεν οι ε, συνθήκες Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν το άρθρο 50 για να φύγει κανείς ε, θέλει, όταν θέλει, ενώ η συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο δεν δίνει καμία δυνατότητα αποχώρηση από τον backstop και θεωρούν ότι δεν σέβεται και τους πολίτες της Βόρειας Ιλλανδίας που είναι υπέρ της Ένωσης τη συνέχιση της ένωσής τους με το Ηνωμένο Βασίλειο. Και θεωρούν, και μου το λένε, ότι δεν χρειάζεται καθόλου backstop. Εφόσον ο Ιρλανδός Πρωθυπουργός είπε ότι δεν θα υπάρξουν σκληρά σύνορα εάν δεν υπάρξει αποχώρηση με συμφωνία. Πολλοί λοιπόν ε, στην Βρετανική Βουλή που πολλοί τους θεωρούν και μετριοπαθείς ε, θεωρούν ότι η έλλειψη συμφωνία είναι καλύτερη από μια κακή συμφωνία. Όμως είδαμε και ότι το εργατικό κόμμα αξιοποιεί οποιαδήποτε ευκαιρία για να δημιουργήσει δυσκολίες στην κυβέρνηση. Ήδη έκαναν πρόταση μομφής και άλλοι πολιτικοί θεωρούν ότι το Κοινοβούλιο ναι μεν ψήφισε υπέρ του Brexit χωρίς να κατανοεί ποιες είναι οι επιπτώσεις του. Θεωρούν λοιπόν ότι μπορούν να αντιστρέψουν το αποτέλεσμα της ε, ε, του δημοψήφισματος αυτού. Είμαστε σε μια κρίσιμη φάση διαδικασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ε, πολύ υπομονητική. Αλλά θα χρειαστεί να περιμένετε λίγο περισσότερο. Πρώτα απ' όλα να δούμε τι θα γίνει με την ε, πρόταση εμπιστοσύνη που πιστεύω θα την κερδίσει. Και κατόπιν η Πρωθυπουργό θα κάνει συζητήσει με όλα τα άλλα πολιτικά κόμματα για να βρει συμφωνία. Άρα έχετε μία επιλογή. Μπορείτε να μην κάνετε τίποτα, να προετοιμαστείτε για την έλλειψη συμφωνία. Μπορείτε να θεωρήσετε ότι μπορεί να σταματήσει το Brexit ή να, να αντιμετωπίσετε μερικέ από τι ανησυχίε των Βρετανών. Για παράδειγμα, να εξηγήσετε στον Ηνωμένο Βασίλειο ότι δεν θέλετε να του κρατήσετε για πάντα στην Ελληνική Ένωση και το backstop θα είναι προσωρινό. Καταλαβαίνω ότι ε, μπορεί να σα φαίνεται ότι σα ζητάω πολλά, γιατί θεωρείτε ότι είναι καλή συμφωνία που προσφέρετε στον Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά όπω και το 2015, όπου εάν είχαν γίνει κάποιε μικροαλλαγέ στι ε, διαπραγματεύσει με τον David Cameron, μπορεί να είχαμε αλλάξει το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματο, νομίζω ήταν πραγματικά κρίμα αν δεν κάνετε περαιτέρω προσπάθειε για να καταλήξουμε σε συμφωνία που θα βοηθήσει τη Βρετανίδα Πρωθυπουργό να φτιάξει, ε, να δημορφώσει πλειοψηφία στο Westminster. Θέλουμε κυρίω ε, αυτό που μα ενδιαφέρει να, είναι, να εστιάζουμε στου πολίτε. Οι αποφάσει μα τι επόμενε μέρε και εβδομάδε θα επηρεάσουν τι δουλειέ, τι επιχειρήσει, την ανάπτυξη τη οικονομία μα. Η επιστολή τη Δευτέρα από του Προέδρου Τούσκ ε, και Γιούνκερ ε, έκανε κάποιε νήξει για περαιτέρω ευελιξία. Α ελπίσουμε ότι αυτή η ευελιξία μπορεί να μεταφραστεί σε συγκεκριμένε προτάσει για να αντιμετωπίσουμε τι ε, ανησυχίε που οδήγησαν στο αποτέλεσμα τη χθεσινή ψηφοφορία. Μόνο τότε θα σταματήσουμε να κοιτάζουμε το παρελθόν και θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε μια πιο ειλικρινή σχέση για το μέλλον. Για τους Ευρωπαίους Φιλελεύθερους και Δημοκράτες, ο κ. Ευχαριστώ πολύ. Θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Είχαμε ελπίσει ένα άλλο αποτέλεσμα, αλλά ε, βλέπουμε τώρα ότι αυτό είναι το αποτέλεσμα της ε, ψηφοφορίας και στην Μεγάλη ε, Βρετανία ε, δεν είχε ήδη μια άποψη σχετικά με το αποτέλεσμα και το τι θα συνέβαινε. Θα πρέπει να σας πω ειλικρινά, δεν έχω εκπλαγεί διότι από το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος είδαμε τι γίνεται στο Whitehall, τις επενδύσεις και είχαμε πάντοτε πλειοψηφίες εναντίον, εναντίον ε, της ιδιότητας του μέλους ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Τελωνιακή Ένωση στην ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων, το Ιρλανδικό ε, backstop και ο κατάλογος είναι πολύ μακρύς. Στη συζήτηση σήμερα το πρωί, κύριε Καμάλ, το ερώτημα είναι πώς να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο και ήλπιζα ότι θα μας δίνατε μια ένδειξη στην παρέμβασή σας. Περιγράψατε την κατάσταση, παρακολουθούμε, αλλά πώς θα βγούμε από αυτό το αδιέξοδο, πώς θα αποφύγουμε το καταστροφικό no deal αυτό το σενάριο και νομίζω ότι η απάντησή μου και νομίζω ότι θα συμφωνείτε μαζί μου χρειαζόμαστε μια μεγάλη πλειοψηφία υπέρ κάποιου, κάποιας λύσης στην Βουλή των Κοινοτήτων και στην Βρετανική πολιτική. Μια πλειοψηφία προς όφελος της Ένωσης και της Βρετανίας μπορούν να επιτευχθούν εάν τα πολιτικά κόμματα, όλα τα πολιτικά κόμματα στη Βρετανία, όχι μόνο το συντηρητικό, αν τα πολιτικά κόμματα αρχίζουν να βάζουν τα συμφέροντα του λαού και της Βρετανίας υπεράνω των στενών κομματικών συμφερόντων. Ας ε, το πω διαφορετικά. Ο κύριος Τζέρεμι Κόμπεν θέλει να γίνει πρωθυπουργός αυτής της χώρας. Η κυρία Μέη ε, θέλει να παραμείνει. Ε, βεβαίως είναι νόμιμο. Ομνόμιμα όλα αυτά αλλά μερικοί θέλουν να χρησιμοποιήσουν αυτό για μια ανεξάρτητη σκοτία. Είναι νόμιμα ότι θέλει να διατηρηθεί η ενότητα της χώρας. Όλα αυτά είναι νόμιμα. Αυτές οι νόμιμες φιλοδοξίες που έχουν όλες είναι όλες νόμιμες. Αλλά αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι ότι το αποτέλεσμα τώρα ε, θα πρέπει να έχουμε ένα σύστημα που να τα υπερβαίνει όλα αυτά. Ένα σύστημα ε, που ε, υπεράνω του συστήματος που παρήγει ανταγωνισμό ανταγωνισμούς. Βεβαίως υπάρχει μια, ένας ανταγωνισμός στο Συντηρητικό Κόμμα ε, στην πλάτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην αρχή της συζήτησης. Σήμερα έχουμε κάτι διαφορετικό. Δεν πρόκειται για μια ε, μάχη μέσα στο κόμμα. Είναι πρόβλημα υπαρξιακό της Βρετανίας, του μέλλοντος της ε, Βρετανίας. Της, δεν, δεν πρόκειται πια για μια μάχη. Εγώ βεβαίως ένας ταπεινός Βέλγος δεν θα κάνω μάθημα ε, στους Βρετανούς ε, για το τι πρέπει να κάνουν, αλλά, αλλά πιστεύω ότι ήρθε η στιγμή να πούμε στους Βρετανούς φίλους μας ότι για το καλό της Βρετανίας θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των κομμάτων στη Μεγάλη Βρετανία όπως το κάνουμε εδώ στο Κοινοβούλιο από την πρώτη μέρα να δούμε ποιες θα είναι οι σχέσεις ανάμεσα στους δύο, να προσδιορίσουμε τις σχέσεις, να βρούμε τις κόκκινες γραμμές ε, που υπήρχαν από την αρχή Βεβαίω, νομίζω ότι σκληρή γραμμή είναι στο συντηρητικό σώμα και εμείς από την Ευρωπαϊκή Ένωση σας λέμε ότι είμαστε έτοιμοι ε, για μια βαθύτερη μελλοντική σχέση, πιο βαθύτερη από ό,τι προβλέπετε. Μισελ στην ε, δήλωση ε, και που επιβεβαιώθηκε πριν λίγα λεπτά και αν υπάρχει στην Βουλή των Κοινοτήτων μια διακομματική πλειοψηφία για μια βαθύτερη τέτοια σχέση, είμαστε έτοιμοι να δεσμευθούμε για να συμβεί αυτό. Υπάρχουν ε, δύο μικρές ανησυχίες. Πρώτα απ' όλα δεν πρέπει να υπάρξει ένα no deal. Είναι επίμαχο αυτό το θέμα ε, και για την ευρωπαϊκή πολιτική καταλαβαίνουμε ότι χρειάζεστε περισσότερο χρόνο. Βεβαίως είναι κακή μέρα ε, να πάμε πέραν του άρθρου 50, ε, πέραν της ημέρας των ευρωεκλογών. Αυτό θα συνεχίσει την αβεβαιότητα για όλους τις επιχειρήσεις. Και δεύτερη ανησυχία είναι το συμφέρον των πελατών, των πελατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασίλου. Deal ή μη deal θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ούτω ώστε να διαφυλάξουμε τα δικαιώματα τους, τα δικαιώματα που υπάρχουν στη Συμφωνία Αποχώρησης με την Επιτροπή ΛΥΜΠ ε, θα ασχοληθούμε με το Βουλή των Κοινοτήτων, με την Επιτροπή τους για να εξασφαλίσουμε τα δικαιώματα, διότι νομίζω ότι όλοι οι πολίτες δεν θα πρέπει ποτέ, ποτέ να είναι τα θύματα των ε, πολιτικών και κομματικών ε, παιχνιδιών, όπως βλέπουμε σήμερα με τον Brexit. Ευχαριστώ πολύ. για την ομάδα των Πρασίνων ο κύριος Λάμπερτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Αυτό που είδαμε ε, χτες ήταν ένας συνασπισμός απίθανος μελών του Βρετανικού ε, Κοινοβουλίου που ψήφισαν μαζικά κατά ενός πράγματος. Αυτό το πράγμα είναι, αν θέλετε, μια ε, συμφωνία η οποία έλαβε, λάμβανε υπόψη τους περιορισμούς τους νομικούς ε, του Good Friday Agreement. Η κόκκινη γραμμή της Βρετανικής κυβέρνησης αυτή καθεαυτή. Είδαμε ότι ε, προσπαθούμε ε, να διαφυλάξουμε την ακεραιότητα και τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό οδηγεί σε τη μόνη δυνατή συμφωνία και εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζουμε στεναρά αυτήν την συμφωνία που παρουσίασε ο Μισελ. Δεύτερο σημείο. Βλέπω ότι ε, μια τροπολογία που κατατέθηκε που ήταν για την δημιουργία μιας δυνατότητας για το Ηνωμένο Βασίλειο μονομερός να βγει από το Good Friday Agreement απορρίφθηκε. Αυτό με ενθαρρύνει. Βλέπω ότι από τις δύο πλευρές της μάχης υπάρχει αποφασιστικότητα να διαφυλαχθεί αυτή η συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής και μην υποτιμάτε τις δυνατότητες που μια δράση μονομερής θα μπορούσε να οδηγήσει και στην Ιρλανδία σε ε, βία. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια μεγάλη πλειοψηφία υπέρ ενός no deal σενάριο. Ένα τέτοιο σενάριο είναι αυτό που αυτόματα ε, λόγω ελλείψεως άλλου θα συμβεί αν δεν υπάρχει πλειοψηφία θετική για μια εναλλακτική λύση. Μια εναλλακτική λύση που θα απαιτήσει από τις αρχές της Μεγάλης Βρετανίας να αναθεωρήσουν τις προσδοκίες τους για μια μελλοντική σχέση. Αντιβουλή των Κοινοτήτων είναι είτε πρόθυμη ή ανίκανη να βρει μια τέτοια θετική πλειοψηφία τότε ως δημοκράτης πιστεύω ότι η μόνη εναλλακτική θα είναι τότε να ζητήσουμε από το Βρετανικό λαό να επιλέξει αν θέλει το Brexit σύμφωνα με τις γραμμές που διαπραγματεύτηκαν τόσο η Βρετανική κυβέρνηση ναι, έτσι καταλαβαίνω τις βρετανικές παραδόσεις ως φιλοφρόνηση και fair play. Ε, νομίζω ότι ε, είχα αρκετό μερίδιο ε, παρέμβασης των ομιλιών μου από τους βουλευτές τους Βρετανούς. Θα ήθελα να δείξουν προσήλωση στις παραδόσεις τους. Γι' αυτό θα ήθελα να παραμείνει το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι μπορείτε να προσφέρετε πολλά στην Ένωσή μας. Νομίζω ότι θα πρέπει ίσως να αποφασίσει ο Βρετανικός λαός μεταξύ του Brexit έτσι όπως έχει ε, συμφωνηθεί η ε, νέα επιλογή. Νομίζω δεν λέχθηκαν πολλά για την οικονομία, της επιχειρήσεις. Θα ήθελα όλοι μας από τις δύο πλευρές της μάχης να λάβουν υπόψη τους 3 εκατομμύρια πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο και 2 εκατομμύρια των Βρετανών που βρίσκονται από αυτή την πλευρά, διότι αυτοί είναι όμοιροι ε, με αυτή την κατάσταση και θα πρέπει αυτό να μας υπενθυμίσει ότι η δημοκρατία και η πολιτική πρέπει να να αναφέρεται κυρίως στην ευημερία και την ευζοία των πολιτών μας. Για την ενιαία Ευρωπαϊκή Αριστερά το λόγο έχει η κυρία Άντερσον. Υποστηρίζουμε εμείς τον backstop γιατί είναι ο λιγότερο βλαπτικός τρόπος για να συνεχίσουμε, αλλά δεν πρέπει να αποδυναμωθεί, δεν πρέπει να γίνει νέα διαπραγμάτευση. Καθημερινά η Βρετανική κυβέρνηση περιφρονεί τον λαό της Ιρλανδίας και αγνοεί τις προβλέψεις της Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής. Το τμήμα του Βρετανικού κατεστημένου, το οποίο υποστηρίζεται από τον DUP, πάντα ήταν εναντίον της συμφωνίας αυτήν. Κάποιοι θεωρούν ότι το Brexit είναι μια καλή ευκαιρία για να απαλλαγούν από τη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής. Δεν υπήρξε ποτέ θετική λύση για την Ιρλανδία από τη Βρετανική Βουλή. Ποτέ στο παρελθόν και ποτέ δεν θα υπάρξει και στο μέλλον. Αυτά τα παιχνίδια, τα απαράδεκτα στο Westminster ε, συνεχίζονται ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να υποστηρίζει τη συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής και υπάρχει κάτι στη συμφωνία αυτή που δίνει μια λύση, δίνει μια διέξοδο και κύριε Φερχώστατη είναι και νόμιμη και δημοκρατική. Λέγει ότι αυτή τη στιγμή ο Υπουργό Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου θεωρεί ότι έχουν υπάρξει αποδείξιμε αλλαγέ σε επίπεδο νοοτροπιών και στάσεων θα προκαλέσει ένα δημοψήφισμα για την Ιρλανδική ενότητα. Έχει υπάρξει τέτοια απόδειξη αλλαγής. Το γνωρίζει η Τερέζα Μέη, το είπε δημόσια, το γνωρίζει η Κάριν Μπράντλεϊ. Η, ε, η Ιρλανδική κυβέρνηση πρέπει να λάβει υπόψη περισσότερο τη δήλωση του Συμβουλίου του Απριλίου 17 το οποίο λέει ότι σε περίπτωση που υπάρξει μια επιτυχής ψηφοφορία επί της Ιρλανδικής Ενότητας, τότε ο, ο τη της Ιρλανδίας θα παραμείνει τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν τω μεταξύ η Ιρλανδία έχει ανάγκη από έκτακτα μέτρα έτσι ώστε να γίνει σεβαστή συμφωνία στο σύνολό της, η συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής. Θα πρέπει να προετοιμαστούμε και να στηρίξουμε τη διεξαγωγή ενός δημοψηφίσματος για την Ιρλανδική Ενότητα. Έχουμε λοιπόν το δικαίωμα να αποφασίζουμε για το μέλλον μας χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις. Αυτό το προβλέπει η Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής. Να προσπαθήσουμε λοιπόν να καθορίσουμε την ένωση στην οποία θέλουμε να ανήκουμε. Ο James Κόνολι έχουν μεγαλύτερη σημασία κάθε μέρα. Είπε ότι η Βρετανική κυβέρνηση δεν έχει κανένα δικαίωμα στην Ιρλανδία. Δεν είχε κανένα δικαίωμα στην Ιρλανδία και δεν θα έχει ποτέ κανένα δικαίωμα στην Ιρλανδία για την Ένωση για την Ελευθερία και την Άμεση Δημοκρατία, ο κύριος Φαράζ. Εξοχότατε κύριε Μπάγνιε, εξοχότατε κύριε Τίμερμαντς. Αυτή είναι η όρη που χρησιμοποίησε η Βρετανή η Πρωθυπουργό ε, στην επιστολή επαιτία που έστειλε πριν ε, από μερικέ μέρε. Αξιοποίησε αυτού του όρου και αυτό είναι απόλυτα συνεπέ με όλη τη διαπραγμάτευση που έκανε. Κατάλαβα στι 8 Δεκεμβρίου του 2017 που θα πήγαινε αυτή η διαδικασία για να τηρήσουμε μια προθεσμία που είχε θέσει ο κύριο Μπάγνιε ο οποίο είναι ένα μη εκλεγμένο γραφειοκράτη των Βρυξελών, η κυβέρνηση, ε, συγγνώμη, η πρωθυπουργό, έφυγε στι 4 πατέρα το πρωί για να σα βρει και υπέγραψε την αρχή του Ιρλανδικού backstop. Είχε πουληθεί η κατάσταση από τότε. Από τότε δεν έχουμε καμία ηγεσία. Και ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι δεν έμαθε το ιστορικό λάθος, δεν έμαθε το ε, ιστορικό δίδαγμα ότι όταν υποκύπτεις αυτούς που σε απειλούν τότε θα σε απειλήσουν ακόμη περισσότερο. Το κείμενο αυτό ήταν ένα κείμενο παράδοσης και το έσκησε χθε η Βουλή των Κοινοτήτων. Είναι σαφές από ό,τι είπατε ότι δεν θα κάνετε περαιτέρω παραχωρήσεις όπως αυτή περιμένει, αλλά εξακολουθεί να είναι πρωθυπουργό μας. Και αυτό από μόνο του είναι αξιοσημείωτο. Αν είχε αίσθηση τιμής θα είχε φύγει τουλάχιστον θα, θα έπρεπε να έχει φύγει μέχρι σήμερα το μεσημέρι. Ορισμένοι λένε ότι κύριε Μπαρνιέ, ε, μα στην ουσία σπαταλήσατε δύο χρόνια τη ζωή σα. Δεν ισχύει αυτό γιατί νομίζω ότι πραγματικά τα φέρατε τα πράγματα όπω θέλατε. Και παρά το ότι 500 ε, βουλευτές ψήφισαν υπέρ του άρθρου 50. Αυτό αποδεικνύει ότι θα πρέπει μετά από δύο χρόνια ή να έχουμε μία ε, συμφωνία ή απλώ να σηκωθούμε να φύγουμε. Και αυτό το λέει και η συμφωνία αποχώρηση του Βρετανικού Κοινοβουλίου που λέει ότι θα φύγουμε χωρί όρου στι 29 Μαρτίου. Αλλά βέβαια εσεί λέτε ότι δεν υπάρχει στήριξη για έλλειψη συμφωνία. Αλλά νομίζατε ότι δεν υπήρχε στήριξη για τον Brexit. Μπορεί να εκπλαγείτε για το πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει η κοινή γνώμη. Κύριε Τίμερμαντ, λέτε ότι αυτό θα κάνει μεγάλη ζημιά αλλά αν ε, όπω ε, είναι νομική μα υποχρέωση αποχωρήσουμε χωρί συμφωνία, θα γίνουμε μια ανεξάρτητη χώρα. Δεν έχει τιμή, δεν έχει τίμημα η ελευθερία. Αλλά παραδέχομαι ότι αμφιβάλλουν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Γιατί βεβαίω ε, στην ουσία τα έχουν βρει μαζί σα. Είναι επίση και ο κύριο Μπλερ και πολλοί άλλοι από το Βρετανικό κατεστημένο που θεωρούν ότι η ψήφο για τον Brexit και γενικά η εκλογή είναι αξιοπεριφρόνητη. Και υπάρχει η θαυμάσια παράδοση. Το είδαμε με τη Δανία, το είδαμε με την Ιρλανδία. Του βάζετε να ξαναψηφίσουν. Τι μπορώ να πω. Αν τελικά καταλήξουμε με παράταση του άρθρου 50, μπορεί να καταλήξουμε να συμμετάσχουμε και στι επόμενε ευρωεκλογέ. Και θα συμμετάσχουμε. Και αν η προδοσία γίνει τέλεια και αν χρειάζεται να κάνουμε δεύτερο δημοψήφισμα, τότε μπορεί να αντιμετωπίσετε μια μεγάλη έκπληξη. Μπορεί να είναι πολύ ήρεμοι και χαλαροί οι Βρετανοί, αλλά άμα του πιέσει, τότε γίνονται λιοντάροι που θα χυμίξει να σα φάει. Θα γίνουν ακόμη πιο ανεξάρτητοι αν γίνει δεύτερο δημοψήφισμα και θα το κερδίσουμε με ακόμη μεγαλύτερη πλειοψηφία. για την ε, ε, ομάδα της Ευρώπης των Εθνών. Για την ομάδα την, ε, για της Ευρώπης των Εθνών και της Ελευθερίας, ο κύριος Μπάτεν. Ευχαριστώ. Εδώ για δυόμιση χρόνια έχουμε καραγκιόζουλίκια. Με βάση λάθο προποθέσει. Ότι δεν μπορεί να φύγει κανεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρί συμφωνία. Μα δεν πρόκειται ποτέ να προκύψει συμφωνία. Δεν θα προκύψει συμφωνία. Η κυρία Μέη και οι διάφοροι απεσταλμένοι του πηγαίνουν προ πίσω, Βρυξέλλε, Λονδίνο, για να καταλήξουν σε μια συμφωνία από χώρε που κανεί δεν τη θέλει. Δεν τη θέλουν αυτοί που θέλουν να παραμείνει, εφόσον δεν θέλουν να φύγει. Δεν τη θέλουν αυτοί που θέλουν να φύγουν, γιατί στην ουσία έτσι δεν φεύγουμε με τέτοια συμφωνία. Και τι εξυπηρετούν όλα αυτά, θα γίνει παράταση, ούτω ώστε τελικά ε, μέσω φθορά ε, να ε, αντιστρέψετε το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματο. Να κουράσετε του εκλογεί. Για πρώτη φορά συμφωνώ με κάτι που λέει ο κ. Φερχόφστατ. Πώ να ξεπεράσουμε το αδιέξοδο στο Βρετανικό Κοινοβούλιο χρειαζόμαστε μια πλειοψηφία υπέρ κάποιου πράγματο. Απόλυτα σωστό, κύριε Φερχόφστατ. Σε τρει μέρε η κυρία Μέη πρέπει να μα υποβάλει ένα δεύτερο σχέδιο, ένα plan B. Υπάρχει ένα plan B που θα έπρεπε να είναι το plan A. Θα ήταν να καταργήσουμε το νόμο του 1972 για τη συμμετοχή στην Ένωση και τότε θα αποχωρήσουμε με βάση του δικού μα όρου και μετά θα δούμε πώ θα καταργήσουμε, θα τροποποιήσουμε με βάση τι δικέ μα προτεραιότητε τι δεκάδε χιλιάδε νομοθετήματα που έχουμε υιοθετήσει έκτοτε. Με το δικό μα χρονοδιάγραμμα. Θα πρέπει να παραιτηθεί αμέσω η κυρία Μέη και να γίνει πρωθυπουργό κάποιο που να θέλει να φύγει το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τη δυνατότητα να αποκαταστήσει την τιμή του. Αν προδώσει το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματο, θα καταστρέψει οποιαδήποτε αξιοπιστία υπάρχει ακόμη για το δημοκρατικό μας σύστημα, που δεν είναι και πολύ υψηλή, αλλά μπορούν να αντιστρέψουν την κατάσταση, μπορούν να πάρουν την πρωτοβουλία, μπορούν να σταματήσουν να σας ζητάνε να του πείτε πώς θα φύγουμε και να αρχίσουμε να λέμε εμείς πώς θα φύγουμε και ο λαό μας ποτέ δεν θα παραδοθεί. κυρία Ντότς, μία εγγεγραμμένη. Ευχαριστώ όσους από την, την Επιτροπή και το Συμβούλιο για τη συνεισφορά τους. Ε, χτες το βράδυ έχουν απορρίψει την ε, συμφωνία. Κάνοντας το αυτό, υποστήριξαν την ακαιρεότητα την ε, συνταγματική θέση της Βόρειας Ιρλανδίας, ε, την ενότητα της ενιαίας αγοράς της Βρετανίας ε, και την προσδοκία για ένα ανεξάρτητο μέλλον εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα το πρωί υπάρχει κάποια σύγχυση σχετικά με την νομική θέση της, Ευρω... της Ηνωμένου Βασιλείου, σχετικά με την παράταση του άρθρου 50 νέου δημοψηφίσματος. Είναι η νομική θέση που θα, από την οποία θα φύγει στις 29 ε, Μαρτίου το Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι σαφές στοιχείο ε, του νόμου. Δεν πρέπει να υπάρχει σύγχυση. Υπάρχει επίσης η πρόταση backstop. Έγινε πολλή λόγος ε, για βία εάν δεν επιτύχει αυτό που θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς στο DUP δεν θέλουμε σκληρά σύνορα. Και Νομίζω ε, ζητώντας ε, το backstop ε, δεν υπάρχει επιλογή no deal επιτάπητος μην επιτρέποντας βιώσιμες αλλαγές, νομίζω έγινε αναπόφευκτο το αποτέλεσμα της χθεσινής ψηφοφορίας. Όλες οι πλευρές είπαν ότι δεν πρέπει να υπάρχουν σκληρά σύνορα με οποιοδήποτε